So, Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ, ας ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολύ φορτωμένο πρόγραμμα και είμαι υποχρεωμένος να ακολουθήσω το χρονοδιάγραμμα. Μάλιστα, υπάρχει και διερμηνία. Στο κανάλι 17, δεν κάνω λάθος, είναι τα ουκρανικά. 25. So, for those following in Ukraine... θέλετε να παρακολουθήσετε την Ουκρανική διερμηνία, το κανάλι είναι το υπαριθμό 25. Κύριε ε, Πρόεδρε της Βουλής Γκρόισμαν, κύριε Αντιπρόεδρε, μέλη Τη Βέρχοβνα Ράντα τη Ουκρανική Βουλή, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, ε, νιώθω ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση για την ευκαιρία που μα δίνεται να βρεθούμε σήμερα το απόγευμα. Δεν είναι αυτά τα επίσημα εγγένεια, είναι μια προκαταρκτική ενημέρωση που οργανώσαμε για να σα δώσουμε μια ιδέα ε, του περιεχομένου τη τη τη ε, αποστολή εκτίμηση αναγκών. Μάλιστα αργότερα το απόγευμα θα σα δώσουμε και αντίγραφο της έκθεσης στα αγγλικά και στα ουκρανικά όταν θα γίνει επίσημη παρουσίαση του εγγράφου στον πρόεδρο της Βουλής, ε, της Ουκρανικής Βουλής, τον κύριο Κρόισμαν και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Σούλτς. Και μάλιστα η ενημέρωση που θα σας κάνω έγινε και χθε προκατακτικά και ε, κατηδίαν από αυρότητα στον πρόεδρο, αντιπρόεδρο και στους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων. Σήμερα δεν πρόκειται να δείξω καμία ιδιαίτερη ευρηματικότητα. Θα επαναλάβω απλώς αυτά που είπα χθε ε, το απόγευμα, ε, ώστε να έχετε όλοι ταυτόχρονα το ίδιο υλικό. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη διαφάνεια. Δεν ξέρω αν μπορείτε να διαβάσετε την οθόνη πίσω μου, αλλά ας δούμε λίγο το ιστορικό. Η Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ Ουκρανίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης ακυρώθηκε ταυτόχρονα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη Βέρχοβνα Ράντα, την Ουκρανική Βουλή, στις 16 Σεπτεμβρίου του 2014. Μάλιστα, είναι μοναδική σημασία σε αυτό το δείγμα και το σημάδι αλληλεγγύης. Γιατί ουδέποτε στο παρελθόν είναι πρωτοφανές ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, μια συνδεδεμένη χώρα να κάνουν αυτή τη χειρονομία, αυτή την αμοιβαία χειρονομία και μάλιστα ταυτόχρονα, με μια ταυτόχρονη κύρωση. Ήταν πρωτόγνωρη αυτή η εμπειρία και δείχνει από την αρχή δίνει το στίγμα της ποιότητας της ιδιαίτερης σχέσης που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ουκρανική Βουλή τη Βέρχοβνα Ράντα. Επόμενη διαφάνεια. Μετά την ομάδα στήριξη δημοκρατίας και συντονισμού των εκλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιλέξαμε την Ουκρανία ως χώρα προτεραιότητας για κοινοβουλευτική δημιουργία ικανοτήτων και διευκόλυνση του διαλόγου. Και πάλι να σας δώσουμε το ιστορικό υπόβαθρο. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας παρατήρησης ε, των βουλευτικών εκλογών ήταν ο Αντρέι Πλέγκοβιτς, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μετά από κάθε εκλογές, ε, οι περισσότερες ε, αποστολές παρατήρησης υποβάλλουν κάποιες συστάσεις. Βέβαια, γενικώ δεν υπήρχε σύστημα παρακολούθησης και κάποιες συνέχειες στην περίπτωση της Ουκρανίας αποφασίσαμε να εξασφαλίσουμε ένα follow-up αναδεικνύοντας τις, τη δέσμευσή μας για συνεργασία με την Βέρχοβνα Ράντα ως προτεραιότητα. Έτσι στις 3 Ιουλίου πέρυσι στο Κίεβο συνυπογράφηκε ένα μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ του Προέδρου Σούλτς, του πρώτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Προέδρου της Ουκρανικής Βουλής, του κ. Γκρόισμαν. Και περνάμε στην επόμενη διαφάνεια. Μετά το Μνημόνιο Συνεννόησης ε, συγκροτήθηκε και μία αποστολή εκτίμησης των αναγκών με μέλη και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη Βέρχοβνα Ράντα για να αναζητηθούν τομείς για ενίσχυση ε, της Βέρχοβνα του δημοκρατικού θεσμού. Και μάλιστα ε, ήταν ιδιαίτερο προνόμιο για μένα που και οι δύο πλευρές του μνημονίου με διόρισαν επικεφαλής της ε, αποστολής αυτής εκτίμησης ε, των αναγκών εκ μέρου και των δύο θεσμικών οργάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ουκρανικής Βουλής. Για να σας πω δύο λόγια για τη μεθοδολογία. Το Σεπτέμβριο του 2016 ε, έκανα μια διερευνητική αποστολή, 2015 μάλλον ο κ. Κόξ, συναντήθηκα με τον πρόεδρο, αντιπρόεδρο, πολλούς αρχηγούς κομμάτων και πολλούς βουλευτές για να προσπαθήσω να καταλάβω ποιο ήταν κατά τη γνώμη των ε, βουλευτών της Ουκρανίας ε, το περιεχόμενο της αποστολής μας. Και έκτοτε είχαμε έξι τέτοιες διερευνητικές αποστολές, ε, πολύήμερες, τριήμερες, τετραήμερες και μάλιστα είχαμε και συναντήσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο πέραν των επισκέψεων και αποστολών και στο Κίεβο. Είχαμε πάνω από 100 συναντήσεις, συνεδριάσεις στο Κίεβο και όλοι όσοι παραγράφησαν σε εκείνες τις ε, συνεδριάσεις ε, και βουλευτές και διοικητικοί, ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, οι οργανώσεις διεθνών φορέων, όλοι, σε όλους μάλλον τρέφουν μεγάλο θαυμασμό και ευγνωμοσύνη. Είχαμε επίσης επίσκεψη και σε διάφορες επιτροπές και μπορέσαμε να συζητήσουμε με τη γραμματεία για να δημιουργήσουμε ε, κάποιες εντυπώσεις για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τελικά εντοπίσαμε 7 συγκεκριμένους τομείς που, θα που θεωρήσαμε ως μοχλούς για μεταμόρφωση, για, για μεταρρύθμιση και σε αυτούς θα επικεντρωθώ. Επίσης, ε, κάναμε και μία επισκόπηση της βιβλιογραφίας, ανάλυση των ε, εγγράφων, γιατί πολλά αναφέρθηκαν για τη Βερχοβνα Ράντα και από επιστήμονες και από πολλές οργανώσεις κοινωνία των πολιτών και της Ουκρανίας. Όλα αυτά τα εξετάσαμε για να δημορφώσουμε μια καλύτερη γνώμη για το τι, ποιο θα ήταν το έργο μα. Και ω προ τη μεθοδολογία θα μπορούσα να πω ότι η αποστολή μας ήταν σαν σφουγγάρι που ρούφηξε κάθε πληροφορία που μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε. Και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα απάβγασμα από όλες αυτές τις πληροφορίες. Αυτή ήταν ουσιαστικά η μεθοδολογία μας. Και περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Για να σας περιγράψω αυτό που ακολουθεί, ε, ήταν σημαντικό να κάνουμε μια, μια μικρή επισκόπηση, γιατί η βασική φιλοσοφία που διέπει την αποστολή είναι η πεποίθηση που εκφράζω και εδώ σήμερα, ότι το μέλλον της Ουκρανίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δημιουργία των θεσμών της. Η αλήθεια είναι ότι παντού στην πολιτική, και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε πολύ ισχυρέ προσωπικότητες. Και μάλιστα ούτε και εσείς ε, έχετε καμία έλλειψη ισχυρών προσωπικότητων στην Ουκρανική πολιτική. Αλλά σε, στο μετασοβιετικό χώρο έχουμε συνδυασμό δυστυχώς ισχυρών προσωπικότητων με ασθενείς θεσμούς. Και αυτό είναι το μήνυμα που θα θέλαμε να στείλουμε, ότι οι θεσμοί πάνω απ' όλα θα πρέπει να, τον, να τονωθούν να δημιουργήσουμε ανεξάρτητους, ισχυρούς, ικανούς και σύγχρονους θεσμούς. Έτσι θα καταφέρει η Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες προκλήσεις. Πώς λοιπόν θα φτιάξουμε ισχυρότερους θεσμούς. Καλύτερα να ξεκινήσουμε από το δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβούλιο της Ουκρανίας και φυσικά καλύτερα να ξεκινήσουμε από τους ερετούς, από τους εκπροσώπους του Ουκρανικού λαού. Αυτή είναι η φιλοσοφία που διέπει την έκθεση. Και μάλιστα οι 7 μοχλοί αλλαγή, οι 7 άξονες αλλαγή που εξετάσαμε είναι η νομοθετική διαδικασία, η νομοπαρασκευαστική διαδικασία ή η νομοθετική εξουσία του Κοινοβουλίου. Αφιερώσαμε πολύ χρόνο στη διαδικασία αυτή τη Ουκρανική Βουλή, τη Βέρχοβνα Ράντα. Τα κοινοβούλια έχουν ευθύνη και κοινοβουλευτική εποπτεία και ελέγχου τη εκτελεστική εξουσία, Στη δική σα περίπτωση, με το σύστημά σας, το προεδρικό, πρωθυπουργικό και διακυβέρνηση, διακυβέρνησης είναι περίπλοκη αυτή η διαδικασία. Το Κοινοβούλιο όμως είναι υπόλογο και προς τους πολίτες. Γι' αυτό χρειάζεται διαφάνεια, άνοιγμα και λογοδοσία προς τους πολίτες. Αυτός είναι βασικός μοχλός. Ε, και μάλιστα με την υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη να θεσπίζει νομοθεσία όπου χρειάζεται και να συνάδει αυτή με την ευρωπαϊκή ένωμη τάξη. Και παρόλο που είμαστε πολιτικοί και ασχολούμαστε κυρίως με τα πολιτικά, ένα πολιτικό σύστημα χρειάζεται και μια σύγχρονη διοίκηση που θα συνδράμει το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό θα πρέπει και η διοίκηση να είναι σε καλή κατάσταση. Εξετάσαμε λοιπόν εδελεχώς και τις διοικητικές ικανότητες της Ουκρανίας. Επίσης είδαμε τα θέματα συνασπισμού, συμμαχίες ε, και σχέση με την αντιπολίτευση και οι δυνατότητες διαλόγου στη Βέρχοβνα Ράντα. Έχετε ένα σύστημα που πολλά πολιτικά κόμματα κάθε φορά που ε, γίνονται εκλογές διαμορφώνεται ένας νέος συνασπισμός ή ένα νέο κόμμα. Και μερικοί εξασφαλίζουν αυτή τη συνέχεια της κοινοβουλευτικής εμπειρίας αλλά πολλοί, 54% στις τελευταίες βουλευτικές εκλογές, είναι καινούργοι, ναι, εκλεγέντες βουλευτές. Πώς λοιπόν θα δημιουργήσουμε συνένεση σε ένα τόσο ρευστό σύστημα. Και οι μέθοδοι μας και τα συστήματά μας μπορούν να βοηθήσουν. Και άλλος σημαντικός μοχλός ε, της ε, μεταρρύθμισης είναι η ηθική ιδεοντολογία και ο κώδικας συμπεριφορά. Οπότε σε 7 άξονες, σε 7 κατηγορίες θα διαπιστώσετε ότι έχουμε συντάξει 52 συστάσεις και 20 από αυτές τις συστάσεις θα σας τις παρουσιάσω σήμερα. Όχι γιατί οι υπόλοιπε 32 είναι ασήμαντες ή λιγότερο ουσιώδεις, αλλά δεν θα, προλάβαμε, θα προλαβαίναμε να ασχοληθούμε με όλες λεπτομεριακά. Θα σας ε, δώσω μια μικρή πρόγευση, θα πάρετε ένα μεζέ κατά κάποιο τρόπο και ελπίζω να έχετε την ευκαιρία αργότερα να δοκιμάσετε ολόκληρο το μενού μας. Ποιε είναι οι 20 βασικέ συστάσει. Ο πρώτο άξονα είναι η νομοθετική, νομοπαρασκευαστική διαδικασία και η νομοθετική ικανότητα τη Βέρχοβνα Ράντα. Η πρώτη μα σύσταση λοιπόν είναι ότι πιστεύουμε πως η Ουκρανική Βουλή και η Ουκρανική Κυβέρνηση και η Προεδρική σα Διοίκηση, Διακυβέρνηση θα πρέπει να συνεργαστούν καθ' όλη τη διάρκεια τη ε, νομοθετική αιτία. Και Δυστυχώς πολλά συμβαίνουν ε, πολύ συχνά, πολύ αργά και με ελάχιστο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται επειδή η όλη η διαδικασία λειτουργεί με τον τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει αν δεν συνεργάζεστε στα διάφορα επίπεδα των θεσμικών οργάνων για να υλοποιήσετε τις αλλαγές που χρειάζονται. Γι' αυτό και επιμένουμε στην ανάγκη να έχουμε ποιότητα του δημοπαρασκευαστικού έργου καθ' όλη τη διάρκεια τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία. Και κάτι άλλο που δεν είναι καινούργιο για το κάνατε και στο παρελθόν, αλλά είναι κάτι που έχει παραμεριστεί. Πριν την κατάσταση από την κυβέρνηση σημαντικών νομοσχεδίων, καλό θα είναι να έχει γίνει μια προκατακτική συζήτηση ενός είδου λευκής βίβλου ώστε να ξέρετε ποιε είναι οι προθέσει, ποιοι είναι οι στόχοι, ποια είναι τα εργαλεία, οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν, το προβλεπόμενο κόστο, οι συνέπειε που αναμένονται. Και μετά να κατατεθεί το νομοσχέδιο στο Κοινοβούλιο, στι Επιτροπέ, στην Ολομέλεια τη Βουλή και να γίνει ένα ψήφισμα, να πει η Βουλή αυτό μας αρέσει, εκείνο δεν μας αρέσει, προτείνουμε κάτι διαφορετικό και πριν γίνει κάτι τέτοιο να συμπεριλάβετε στι διαβουλεύσει και την κοινωνία των πολιτών, εμπειρογνώμονες από την παιδεία, την ε, υγεία, την γεωργία, την ευημερία για να γίνεται ε, μια πραγματικά ζωντανή Βουλή, να γίνεται ο παλμός της κοινωνίας, της Ουκρανικής κοινωνίας και να βελτιώσετε έτσι την ποιότητα του έργου σας, ώστε να γίνει το έργο σας ε, το έργο για τους Ουκρανούς πολίτες ε, για το καλό του λαού σας, τον ψηφοφόρο σας, αυτόν που εκπροσωπείτε. Δεν είναι τίποτα φοβερό και καινοτόμο, δεν είναι το τραγωνισμό του κύκλου. Θα πρέπει να αρχίσετε να εργάζεστε για τους Ουκρανούς, για χάρη των Ουκρανών εντός της Ουκρανίας. Επάραμε στην επόμενη διαφάνεια. Ένας από τους τομείς, και μάλιστα δεν θα εκπλαγούν ε, όσοι ήδη έχουν συζητήσει αυτά τα θέματα, ένα που διακρίνει την ε, δική σας βουλή είναι η χρήση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, το δικαίωμα της ε, νομοθετικής πρωτοβουλίας από μεμονωμένους βουλευτές. Αποδεχόμαστε αυτή την ιδιαιτερότητα, αυτό το δικαίωμα, γιατί πολλές βουλές το προβλέπουν. Αυτό όμω που διαφοροποιεί τη Βέρχοβνα Ράτα από τα άλλα κοινοβούλια που έχουν κατοχυρώσει αυτό το δικαίωμα είναι ότι στη δική σας περίπτωση έχουμε τεράστιο όγκο των νομοσχεδίων που εκπορεύονται από τέτοια ιδιωτική πρωτοβουλία βουλευτών. Μάλιστα, μέχρι στιγμή είχατε 2.500 νομοθετικές προτάσεις. 2.000 από αυτές ε, ήταν ε, νομοθετικές πρωτοβουλίες ε, μεμονωμένων βουλευτών. Και ο πρόεδρος, η πρόεδρο των επιτροπών λέμε δεν μπορούμε να χειριστούμε αυτό τον όγκο. Και νομικές υπηρεσίες μας λένε προσπαθούμε να διορθώσουμε τις διατυπώσεις, αλλά είναι τόσο όγκος που όλοι αγχώνονται. Είναι σαν να έχουμε αυτά τα spam που έχουμε στους, ε, ε, στις, ε, στους υπολογιστές, τα ανεπιθύμητα mail που λαμβάνουμε. Είναι σαν ένα παλιριακό νομοθετικό κύμα που κατακλείζει τις υπηρεσίες της Βέρχοβνα Ράντα. Και αυτά είναι στατιστικά στοιχεία που λάβαμε από τη Βέρχο Βεναράδα και διαπιστώσαμε ότι τον ίδιο χρόνο μόνο 7% των προτάσεων μετεξελίχθηκαν σε νομοθέτημα, σε νομοθετικές διατάξεις. Οπότε σκεφτείτε το. Αν εσείς ήσασταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μιας εταιρείας και έρχονταν οι μάνατζερ, οι διοικητικοί διευθυντές και σας έλεγαν Είχαμε 100% της προσπάθειας, αλλά μόνο 7% αποτέλεσμα. Θα ρωτήσετε εύλογα, τι έγινε με το 93%? Μήπως δεν έγινε καλή αξιοποίηση των πόρων? Φαίνεται ότι έγινε κατασπατάληση των πόρων. Αυτό λοιπόν διαρωτόμαστε και εμείς. Γι' αυτό και η σύστασή μας είναι να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των μελών για νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά ο κατάλογος των 2.000 προτάσεων ε, να μειωθεί και μάλιστα κάθε πολιτική ομάδα ανάλογα με το μέγεθός της να μπορεί να επιλέγει. Οπότε, άσχετα αν είναι κανείς κυβερνών κόμμα ή αντιπολίτευση, ανάλογα με το μέγεθός του να έχει ένα μερίδιο ε, των ε, νομοθετικών προτάσεων και να επιλέγει τις 20 προτεραιότητες και μετά να γίνεται και ένας ε, έλεγχος ποιότητας. Σωστή νομοθετική διατύπωση, μελέτη επιπτώσεων, συνάφεια με το Σύνταγμα, συνταγματικότητα, ουδετερότητα, ευθυγράμμιση ε, με το κοινοτικό κεκτημένο. Ήδη τα έχετε όλα αυτά στους κανόνες, αλλά τα γνωρίτε. Οπότε εφαρμόστε τους κανόνες, τους υφιστάμενους κανόνες και μετά πάτε στη Βουλή, στην Ολομέλεια και ψηφίσετε. το. Αν ψηφίσετε σε μία σύνοδο ε, της 20 θα πολλαπλασιαστούν την επόμενη φορά. Γιατί κάθε φορά θα έχετε 20 νέες προτάσεις. Αλλά τουλάχιστον οι επιτροπές σα που θα έχουν πάντα 20 προτάσεις θα απαιτούν καλύτερο διοικητικό έλεγχο από την διοίκηση. Θα προλαβαίνουν να διαβουλεύονται με τους εμπειρογνώμονες και να πηγαίνουν στην Ολομέλεια και να ψηφίσουν υπέρ ή κατά. Και όταν τελειώσει και οταν τελειωσει η ψηφοφορια θα ανανεώνεται ο κατάλογος. Οπότε δεν είναι μόνο 20 συνολικά, είναι 20 κάθε φορά, αλλά τουλάχιστον δεν είναι 2.000. Ένα τέτοιο παλιριακό κύμα νομοθετικό που θα πνίγει στη Βέρχοβνα Ράδα. Θα πρέπει και οι... να βάζουν οι βουλευτές κάποια προτεραιότητα μέσα των κομμάτων τους. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουμε αυτή τη μέθοδο, γιατί δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα ιδιωτική νομοθετική πρωτοβουλία. Αλλά και άλλα κοινοβούλια στην Ευρώπη έχουν αυτό το δικαίωμα. Γι' αυτό σα στείλουμε αυτή τη μεθοδολογία. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε το ημερολόγιο αναμήνα του κοινοβουλευτικού έργου. Πάλι εξετάζουμε τις πληροφορίες. Τα γνωρίζουμε όλα. Όχι, δεν γνωρίζαμε τίποτα, αλλά ρωτήσαμε. Και αυτό που ανακαλύψαμε είναι ότι στην πρακτική που ασκείτε στην Βουλή σας, Βερκόφνα Ράντα, όταν έρχεστε στο Κίεβο για να συμμετάσχετε στις Ολομέλειες, θέλετε στην ίδια εβδομάδα να συνεδριάσουν και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές. Και στη διάρκεια της Ολομέλειας, εβδομάδας της Ολομέλειας, συμμετέχετε και στην κοινοβουλευτική Επιτροπή. Εμείς εξετάσαμε τις πληροφορίες για την εβδομάδα των κοινοβουλευτικών επιτροπών και διαπιστώσαμε ότι στην εβδομάδα που είναι αφιερωμένη στο έργο των κοινοβουλευτικών επιτροπών οι περισσότερες δεν ε, συνεδριάζουν και όσοι συνεδριάζουν δεν έχουν συνήθως απαρτία. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι οι εβδομάδα αυτή που είναι αφιερωμένη στις κοινοβουλευτικές επιτροπές είναι στην ουσία ένα πλάσμα, δηλαδή δεν είναι πραγματικότητα. Και όσους συνάντησα και ιδίω προέδρους κοινοβουλευτικών επιτροπών μου είπαν «Μα δεν έχουμε χρόνο σε επιτροπές μας για να διεκπαιρεώσουμε το έργο μας». Δώστε περισσότερο χρόνο σε αυτούς σας στην Βουλή και κάντε τις εβδομάδες μικτές. Τώρα πόσες θα προσθέσετε είναι δική σας υπόθεση. Όλα βεβαίως είναι δική σας υπόθεση. Η δική σας βουλή είναι, δική σας εντολή είναι και δικό σας σύνταγμα είναι. Η δική μας συμβουλή προς εσάς είναι αν δεν έχετε χρόνο να εργαστείτε, αν δεν έχετε παρκή χρόνο να εργαστείτε τότε δώστε στους αυτούς σας περισσότερο χρόνο. Τώρα στην επόμενη διαφάνεια σας παρακαλώ σχετικά με τη λειτουργία του Συμβουλίου Συνδιαλλαγής για την ε, θέσπιση των εργασιών. Εμείς νομίζουμε ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να αναθεωρηθεί και ότι αυτή, ε, αυτό το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζει και κλεισμένο των θυρών. Θέλω να πω στους εκπροσώπους ε, της κοινωνίας των πολιτών ότι αυτό δεν έχει σκοπό να αποκλείσει ιονδήποτε. Θα δημοσιεύετε την ημερήσια διάταξή σας και θα γνωρίζουν όλοι. Εγώ είχα το προνόμιο ε, να είμαι πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και πρόεδρος πολιτικής ομάδας. Ορισμένα πράγματα σας αναγκάζουν να συνεδριάσετε και κλεισμένο των θυρών αναζητώντας τον δρόμο προς τον οποίο θα κινηθείτε. Όταν όμως θα έχετε αποφασίσει όλοι έχουν το δικαίωμα να μάθουν ποια είναι η αποφασή σας. Ορισμένα από τα πράγματα αυτά είναι βαρετά. Όμως καμιά φορά τα βαρετά πράγματα μπορούν να είναι πάρα πολύ καλά, πολύ θετικά, εφόσον σας επιτρέπουν να αποδώσετε. Και αυτό που διαπιστώσαμε κάποτε όταν πήγαμε στο Συμβούλιο Συνδιαλλαγή και εγώ εξεπλάγει διότι είδα ένα πλήθο ε, τηλεοπτικών συνεργείων. Αυτό που κάνετε όταν έχετε μια σειρά τηλεοπτικών συνεργείων μπροστά σε ένα πολιτικό, ξέρετε τι θα κάνει. Hollywood θα δείτε στην πραγματικότητα. Α, να κερδίσετε το Όσκαρ και επομένως στην ουσία παίζετε ένα ρόλο μπροστά στην κάμερα. Το πρόβλημα όμως όταν το βλέπετε αυτό είναι ότι δεν κάνετε τα βαρετά πράγματα που κάνετε 10 το πρωί την Τετάρτη όταν ψηφίζετε και λαμβάνετε το λόγο κτλ. Καμιά φορά λοιπόν ίσως το χρωστάτε και εσείς στους εαυτούς σας κύριε Πρόεδρε και εσείς Αντιπρόεδρε να κάνετε σωστά και τα βαρετά πράγματα ώστε να λειτουργήσει το σύστημα καλύτερα και τελικά μετά να δώσει το δικαίωμα σε όλους και όλους να γνωρίζουν τι αποφασίζετε. Όσον αφορά το σύστημα ψηφοφόρια σας. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ είναι βέβαια ευαίσθητο θέμα. Εκπλαγήκαμε από το ύψος της απαρτίας σας. Ότι χρειάζεται δηλαδή το μισό των 450 συν 1, δηλαδή 226. Αλλά βέβαια δεν έρχονται από την Κρυμαία, διότι έχει προσαρτηθεί. Όχι από τον Βέσκ, από τον Νιέσκ, γιατί ε, και εκεί είναι γνωστά τα προβλήματα. Έχει, ξεκολουθείτε όμως να έχετε βάλει την απαρτία σας πάρα πολύ ψηλά, παρόλο που σας λείπουν ορισμένοι βουλευτές σας. Εμείς νομίζουμε ότι πρέπει να συνεννοηθείτε, να μειώσετε, να κατεβάσετε τον πύχη για να μπορέσετε να αποδώσετε. Γιατί τι συμβαίνει όταν ο πύχης είναι τόσο υψηλά. Όλοι γνωρίζουμε. Στην ουσία δεν ψηφίζετε και στην ουσία χάνετε την αξιοπιστία σας. Δηλαδή, τι γίνεται ο, ο πρόεδρος ελέγχει και ξαναελέγχει και ξαναελέγχει και ανεβοκατεβαίνει η απαρτία. 219, 220, 222, τα φτάσει 226, τότε πατάτε το κουμπί και ψηφίζετε. Δεν είναι καλός τρόπος. Ορισμένοι λένε ότι θέλετε υψηλό κατόφλιο. Αν θέλετε βεβαίως να αναθεωρήσετε το Σύνταγμα, ασφαλώς και χρειάζεται πολύ υψηλή απαρτία. Είναι σημαντικό κείμενο. Όμως, πολλά νομοσχέδια θα πρέπει να ψηφίζονται με χαμηλότερο κατόφλιο. Στην ομάδα μας συζητήσαμε πολύ σχετικά με το ερώτημα αν θα πρέπει να σας τα πούμε αυτά ή όχι. Εγώ θα σας το πω διότι αυτά είναι και στο Σύνταγμά σας, έτσι. Δεν είναι δική μας αποστολή βεβαίω να αναθεωρήσουμε το Σύνταγμά μας, κανένας δεν μας το ζήτησε αυτό. Το μόνο που σας λέγω εδώ είναι αν θεωρείτε ότι είναι καλό. Αν θεωρείτε, δηλαδή, ας πούμε μια τεχνική τροποποίηση του συντάγματο χωρίς να προκαταλάβετε καθόλου την ε, ουσία αν θα είναι προεδρευόμενη η προεδρική δημοκρατία σας κτλ. Είναι καθαρά τεχνική αλλαγή. Δεν πρόκειται να αλλάξει ε, τα θεμέλια του συστήματος ούτε την ε, μετακύληση των αρμοδιοτήτων κτλ. Νομίζω ότι είναι κάτι που θα σας φανεί χρήσιμο και που είναι και σημαντικό για τον πολιτισμό του κοινοβουλευτισμού. Δηλαδή να ευθυγραμμιστούν οι εργασίες με τις εργασίες άλλων κοινοβουλίων. Φανταστείτε κάποτε να κερδίσει αντιπολίτευση με τον νέο κανόνα. Αυτό για μένα είναι καλό για τη δημοκρατία. Διότι είναι ένα, σήμα αφύπνισης αν θέλετε πραγματικά να πάτε να δουλέψετε. Θα βάλει λοιπόν στο σύστημά σας τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και αλλού το WIP, δηλαδή τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, που επιμένει να είναι παρόντες οι βουλευτές. Αυτό σε επίπεδο νοοτροπίας δεν θα γίνει αν δεν δημιουργήσετε τις προϋποθέσεις για να επιβληθεί. Γι' αυτό σας συνιστούμε πολύ θερμά να το σκεφτείτε παρόλο που ίσω να σα φανεί ότι κάπω υπερβαίνουμε τα όρια τη εντολής μα και δεν θέλουμε καθόλου να σα δώσουμε την εντύπωση ότι εξετάζουμε το σύνταγμά σα. Αυτό είναι μια τελείω διαφορετική συζήτηση στην οποία δεν αναμειχθήκαμε καθόλου. Τώρα, ένα άλλο θέμα σε ό,τι αφορά την πολιτική εποπτεία, τον έλεγχο δηλαδή τη εκτελεστική εξουσία από τη Βουλή. Πάρα πολύ σημαντικό για οποιοδήποτε κοινοβούλιο. Ποιο, πώς ασκείται τον έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία. Θα σα πω κάτι. Ένα παράδειγμα, κάπω ακραίο βέβαια. Το 1998-99 είχαμε ένα μεγάλο καυγά ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλω να σα βαρύνω με διάφορε λεπτομέρειε, αλλά πρόκειται για θέματα λογοδοσία, accountability. Και στο τέλο, για πρώτη φορά και μοναδική, αναγκάστηκε ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρετηθεί. Όχι επειδή ήμασταν κατά τη ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε κατά τη Ευρώπη. Ήταν διότι δεν μας άρεσε η έλλειψη λογοδοσίας διότι αυτό είναι το αίμα που κυκλοφορεί στις αρτηρίες μιας πραγματικής βουλής. Λοιπόν, να το ρυθμίσετε σωστά, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τους πολίτες και για τις κοινοβουλευτικές σας επιτροπές, για την ακερότητα του Κοινοβουλίου, για τον ρόλο του βουλευτού. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι πιστεύουμε ότι η Βερχόφνα Ράντα και ιδίω βεβαίω το Υπουργικό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσετε από κοινού ένα τύπο για τις ετήσιες υποβολές εκθέσεων στη Βερχόφνα Ράντα. Πότε θα αναμένετε να λάβετε τις εκθέσεις αυτές, τι θα τις κάνετε, ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, πότε είναι ουσιώδες να είναι παρόν ο Πρωθυπουργός και πότε όχι. Δεν χρειάζεται και τους υπουργούς άλλωστε κάθε μέρα. Τον χρειάζεται όμω σε σημαντικέ πολιτικά ημέρε. Αυτά όλα θέλουν κάποιο σχεδιασμό και μια κατάλληλη διαδικασία. Θα σα πούμε επίση ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να περιλάβει και αυτό είναι σημαντικό για να ασκήσει σωστά τον εποπτικό του ρόλο το κοινοβούλιο, θα πρέπει να περιλαμβάνει και το σχεδιασμό του περσινού έτους και την έκβαση του σχεδιασμού αυτού, διότι αυτό που σας ενδιαφέρει είναι τελικώς να έχετε κάποια αποτελέσματα. Όχι απλά να δημοσιεύσετε κάποιο νομοθετικό κείμενο, αλλά πώς εφαρμόστηκε εν τέλει. Και αν δεν εφαρμόστηκε, γιατί δεν εφαρμόστηκε. Αυτή είναι η δουλειά του Κοινοβουλίου, να μπει στο γιατί όχι. Συνιστούμε λοιπόν πολύ θερμά να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό. Και στην επόμενη διαφάνεια τώρα, για την πολιτική εποπτεία, εμείς θεωρούμε ότι έχει υπερβολικά πολλές επιτροπές. 28 συν 1 νομίζω για το μέγεθος της Βουλής σας. Δεν θα σας πούμε εμείς βεβαίως πόσες πρέπει να έχετε. Εμείς νομίζουμε πάντως θα πρέπει να είναι λιγότερες. Ιδεοδός θα πρέπει να έχετε μια κοινοβουλευτική επιτροπή που να ελέγχει ένα Υπουργείο, ώστε να γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς λειτουργούν τα πράγματα αυτά. Εξάλλου, συνιστούμε θερμά, ήδη από τώρα, από τούτην εδώ την εντολή, η Βερχόφνα Ράζα να ε, συμφωνήσει επ' αυτού για την επόμενη θητεία. Γιατί το λέω αυτό, γιατί είμαι και άνθρωπος με πρακτικό πνεύμα και από το παρελθόν μου. Σήμερα έχετε προέδρους, αντιπροέδρους και ούτως εξής όλα τα σχετικά αξιώματα. Αν τους διώξετε όλους αυτούς την επόμενη εβδομάδα, τελείωσε. Θα είναι θνησιγενής η πρόταση, διότι ο κόσμος αυτός θα θέλει να κρατήσει τη θέση του. Όμως, θα σχεδιάσετε για το μέλλον. Και αν σχεδιάσετε για το μέλλον, θα μπορέσει να λειτουργήσει, διότι θα είναι μια πρόσω συνένεση, μια συνένεση για το μέλλον. Αυτό που θα, ναι, επόμενη διαφάνεια, θα προτείνουμε είναι να προσθέσετε κάτι ακόμη. Να πείτε δηλαδή ότι θα εξετάσετε το ενδεχόμενο να προσθέσετε την εφαρμογή ενός πράγματος που λέγεται μέθοδος de Hont. Ενός θανόντος τώρα πια ε, Βέλγου στατιστικολόγου. Αυτή η μέθοδος de χρησιμοποιείται σε πολλά κοινοβούλια και, σε, και στο ευρωπαϊκό Δώσαμε χθε σε όλους τους επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών ομάδων ένα σχετικό σημείωμα να πάνε να σπάσουν τα κεφάλια τους όταν θα επιστρέψουν στο Κίεβο, αλλά να συζητήσετε μαζί τους και θα μιλήσουμε και εμείς. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι υπό το σύστημα The Hunt φανταστείτε ότι έχετε 20 κοινοβουλευτικές επιτρόπες και 9 αντιπροσωπείες. Άρα συνολικά έχετε 29 πακέτα, ας πούμε. Το καθένα έχει ένα πρόεδρο, αντιπρόεδρο ή αντιπρόεδρος κλπ. Άρα θα έχετε τρεις φορές 29 θέσεις. Τα βάζετε στο τραπέζι, σαν μια μεγάλη τούρτα. Και το σύστημα τεχών είναι ο τρόπος με τον οποίο θα κόψετε την τούρτα. Σας λέει πόσα κομμάτια από την τούρτα θα λάβετε. Και ο αριθμός των κομματιών της τούρτας έχει σχέση με την αριθμητική σας δύναμη. Οι μεγάλες κοινοβουλευτικές ομάδες, πολύ τούρτα. Μικρές κοινοβουλευτικές ομάδες, λίγο μέρος από την τούρτα. Το σύστημα τεχόντ λέει όμως ποιος θα διαλέξει πρώτος, δεύτερος, τρίτος κλπ. Και ως αποτέλεσμα έχετε εν τέλει ένα σύστημα όπου αν συμφωνήσετε επί της μεθοδολογίας και του αριθμού των επιτροπών, πάει καλά, δεν χρειάζεται όμως να δείτε θα Δηλαδή, θα ξεκινήσετε λέγοντα ότι, μια, ότι συνιστάται μια κοινοβουλευτική επιτροπή έναντι κάθε Υπουργείου. Μετά ναι, αλλά ε, έχουμε και αυτόν τον Κόξ που θέλει τέτοια καλά να αποκτήσει κάποια ε, θέση. Θέλει να είναι κάπου αναπληρωτή. Και θα έρθει κάποιο άλλο. Ναι, μα έχουμε και τούτον εδώ που θέλει επίση μια δουλειά. Α φτιάξουμε άλλη μια επιτροπή. Καταλήγεται τότε να αναστατώνετε ολόκληρο το σύστημα για να αντιμετωπίσετε τι ανάγκε αυτές. Αν μπορείτε να συμφωνήσετε εξ αρχής να ρυθμίσετε τον αριθμό των κοινοβουλευτικών επιτροπών και τον τρόπο επιλογής μπορείτε να έχετε ένα σύστημα που να λειτουργεί και θα έχετε τότε υπουργού που θα εποπτεύονται και θα λογοδοτούν σε μια συγκεκριμένη κοινοβουλευτική επιτροπή. Σα συνιστούμε λοιπόν πολύ θερμά να το μελετήστε το θέμα αυτό. Και μια τελευταία σύσταση, γιατί υπάρχουν και άλλε συστάσει μέσα στο ίδιο το κείμενο. Κάτι δηλαδή που ίσω θα σα ενδιέφερε για να αναπτύξετε τι κοινοβουλευτικέ δεξιότητε είναι το σύστημα των εισηγητών. Σα δείχνω μια μελέτη τη Επιτροπή Προπολογισμών και από το Ινστιτούτο GIZ του ε, Βερολίνου λέει πώ λειτουργεί το σύστημα των εισηγητών για τον προπολογισμό. Εξετάστε το έγγραφο και θα δείτε ποια είναι η ιδέα που είναι να αναπτυχθούν δεξιότητες των κοινοβουλευτικών που βεβαίως θα υποστηρίζονται και από τις δεξιότητες των ε, αξιωματούχων της διοίκησης. Ξέρω ότι φτιάχνατε προϋπολογισμό τελευταία στιγμή. Λόγω της κρίσεως, ναι. Τελευταία μέρα του Δεκεμβρίου. Ναι, αλλά κοίταξα τα τελευταία σας 10 χρόνια και το κάνατε με τον ίδιο τρόπο και πριν από την κρίση. Δεν είναι υπεύθυνο τρόπος και δεν μιλάω εδώ για λαϊκισμό. Μιλώ για την ουσία της αντιμετώπισης αυτών των θεμάτων πολιτικής. Ας έρθω τώρα στο υπαριθμόν 3 που είναι το ανοιχτό πνεύμα η διαφάνεια και η λογοδοσία στους πολίτες. Βεβαίως εδώ και επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες τις τελευταίες εβδομάδες, όποιες έχετε κάνει. Να φτιάξετε μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική, όχι μόνο με τον εξοπλισμό, αλλά και μια νέα ε, νοοτροπία, μια νέα φιλοσοφία και βεβαίως νέες δεξιότητες για το πώ θα τα χειριστείτε αυτά. Το Ευρωπαϊκό Κοινόβουλιο είναι διατεθειμένο να συνεργαστεί με τη Βερχόφνα Ράδα σε μια άνευ προηγουμένου εταιρική σχέση για παροχή συμβουλών, στήριξη και συνεργασίας στην ανάπτυξη της στρατηγική, εάν τελικώς αποφασίσετε ότι τη θέλετε και εμεί σα τη συνιστούμε επίσης πολύ θερμά. Χρειάζονται επαρκή πόροι και είναι και ένας τρόπος να έρθει σε επαφή με πιο σύγχρονο τρόπο η Βουλή με το ευρύ κοινό. Δεν έχετε επαρκή πόρου για την ώρα, πάντω όχι στον προπολογισμό σα για να στηρίξετε προσπάθεια τέτοιου Εύρου. Άρα χρειάζεται να γίνει πολλή δουλειά. Ακόμη και καθώ τώρα που κάνουμε τη σύσταση και να μα πείτε εσεί ναι, χρειάζεται πολλή χρόνο και πολλή δουλειά και προσπάθεια ακόμη μέχρι ότου υλοποιηθεί αυτό το ναι. Πέραν αυτού, αλλάξτε διαφάνεια, να δούμε και μία σε βάθο στρατηγική επικοινωνίας. Ποιο είναι το ακροτηριό σα, ποιο είναι ο προπολογισμό σα, τι είδου στρατηγική διαθέτεται για τον θεσμό σας. Και δεν μιλώ εδώ για την κάθε μια κοινοβουλευτική ομάδα ξεχωριστά. Μιλώ για τον θεσμό της Βερχόφνα Ράντα, η οποία χορηγεί πληροφορίες στους πολίτες. Και βεβαίως για τις κοινοβουλευτικές ομάδες και για την πολιτική που ασκεί ο καθένας. Όμως το σύστημα αυτό θα πρέπει να έχει και μια εύκολη δίωδο ώστε να πηγαίνει για, σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα και μέσα σε κάθε κοινοβουλευτική ομάδα να υπάρχει και ένα σύνδεσμο να σα πάει σε κάθε ένα βουλευτή. Για την ώρα αυτό το σύστημα ίσως να βρίσκεται στον χώρο του ονείρου και όχι στην πραγματικότητα. Γι' αυτό και πρέπει να εγγύψετε στην προσπάθεια αυτή. Έχετε μερικούς πολύ άξιους και ικανούς ανθρώπους και στην τηλεόραση και στα περιοδικά και στι εφημερίδες που γνωρίζουν επικοινωνία. Χρειάζεται να κάνετε μια προσπάθεια να τους προσελκύσετε και πάλι να συνδεθούν με μια κεντρική στρατηγική που θα είναι σχεδιασμένη να εκπροσωπεί τις ανάγκες των βουλευτών του σήμερα και της κοινωνίας του σήμερα. Τώρα μοχλός υπαριθμών 4, προσέγγιση του, της Ουκρανικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εδώ μπορούμε πολλά πράγματα, θα πω ένα μονάχα να έχετε υπόψη σας. Ο νόμος που έχετε σήμερα στην Ουκρανία σχετικά με φιλική προς την Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθεσία είναι πλέον απειρχαιωμένο, διότι χρονολογείται από πριν από την Συμφωνία Συνδέσεως. Άρα πρέπει να γίνει πιο επίκαιρο. Να σηκωθεί ο νόμος να πάει στο σχολείο να μάθει τι γίνεται και να επανέλθει. Όχι μόνο διότι η Συμφωνία Συνδέσεως είναι υψηλότερο επίπεδο συνεργασίας από το προηγούμενο, έρχομαι τώρα στο 5, δηλαδή διοικητικέ ικανότητε νούμερο 5 μεν, αλλά όχι πέμπτο σε ιεραρχία. Αν θέλετε μια βουλή που να αποδίδει έργο πραγματικά, χρειάζεστε ποιοτική διοίκηση. Έχετε μερικούς πάρα πολύ ικανούς αξιωματούχους, έχετε και πολύ ικανούς βουλευτές. Έχετε όμως απειρχιωμένα συστήματα. Άξιος κόσμος με απειρχιωμένα συστήματα δεν αποδίδει. Καλοί αξιωματούχοι και καλά συστήματα αποδίδουν. Σε ό,τι αφορά τη διοίκηση σα κάτι που θα πρέπει να έχετε το δικαίωμα να κάνετε θα είναι να θεσπίζετε εσείς τον δικό σας προπολογισμό. Δεν σημαίνει να σηκωθείτε να πάρετε το 1 τέταρτο από τον ε, ήδη ε, ε, στριμωγμένο προπολογισμό της χώρας σας. Όχι, να διαθέσετε επαρκεί πόρους για να μπορείτε να διοικείτε τη Βουλή σας σωστά. Και εφόσον θα, θα φανείτε λογικοί και οι άλλοι θεσμοί θα σας στηρίξουν σε αυτό. Όμως θα πρέπει να υπάρχει και ένα τίμημα. Αν σας δώσουν περισσότερα πράγματα θα πρέπει να αποδώσετε και εσείς με περισσότερη λογοδοσία. Διότι είναι περιορισμένα τα δημόσια οικονομικά. Εσείς ψηφίσατε υπέρ του νέου ελεγκτικού συνεδρίου και εν πάση περιπτώσει πρέπει να ακούσετε τι λέει. Το λέω αυτό για δύο λόγους. Αφενός η διαφάνεια θα σας αναγκάσει να βάλετε προτεραιότητα στις δαπάνες σας, διότι θα κληθείτε μετά να λογοδοτήσετε για αυτές. Και δεύτερο, το κοινό θα γνωρίζει τι πράτετε και θα μπορεί να αντιδρά και να σας λέει ποια είναι η γνώμη του. Και τρίτο, θα δώσετε και το παράδειγμα και στους άλλους θεσμούς στην Ουκρανία που ίσως να, ίσως να μην θέλουν να έρθει το ελεγκτικό συνέδριο να εξετάσει τι κάνουν αλλά εάν δουν ότι η Βουλή ανοίγει τα βιβλία της, τότε και οι υπόλοιποι θα το δεχτούν. Αυτή είναι η εντολή που σας έδωσε η Μαϊντάν και θα είναι και σωστό παράδειγμα. Φτιάξτε εσείς τον προϋπολογισμό σας, ε, θεσπίστε τα σχετικά με τη λογοδοσία, εμείς θα είμαστε στο πλευρό σας. Νομίζουμε επίσης ότι πρέπει να ενισχύσετε τον πυρήνα της διοίκησής σας. Έχετε πολλούς καλούς ανθρώπους αλλά είναι εκτός. Πήγα να βρω την κοινοβουλευτική σας βιβλιοθήκη και τη βρήκα στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ε, ας είναι και στον Άρη. Πού να πάω να τη βρω. Χρειάζεστε εμπειρία. Έχετε εμπειρία αλλά πρέπει να συνδεχθεί και να έρθει να σας βρει, να την προσελκύσετε για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκε των βουλευτών, των κοινοβουλευτικών επιτροπών κ.ο.κ. Ένα τελευταίο σχόλιο υπό την επικεφαλίδα αυτή πάντα είναι ότι χρειάζεται μια πολιτική ανάπτυξη του προσωπικού, διότι κουβαλάτε ακόμα πολλέ κληρονομιέ του παρελθόντο. Και το ίδιο το όνομα. Δεν μιλώ ουκρανικά βέβαια, αλλά αυτό το απαράτ, ο διοικητικό μηχανισμό δηλαδή και ο απαράτσικ Αυτά τα πράγματα προέρχονται από το παρελθόν. Ό,τι σας λένε κάνετε. Αυτό όμως πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να βρείτε αυτό που λέγεται middle management, η μεσαίη manager και αυτοί να είναι άνθρωποι ικανοί και με προσόντα και να εμφυσίσουν νέα πνοή στην δουλειά αυτή χρησιμοποιώντας και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής με εκπαιδευμένους ανθρώπους, επαγγελματίες Γνωρίζετε ότι σήμερα στη Βερχόφνα Ράντα ο προϋπολογισμός κατά κεφαλήν για την εκπαίδευση είναι περίπου 2,5 ευρώ. Μα αυτό είναι ένας καφές. Ένας καφές στις 11 το πρωί. Δεν είναι πραγματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης. Αν θέλετε να προσφέρετε στους εαυτούς σας ως βουλευτές ένα γερό σύστημα για να σας ενισχύει, να σας υποστηρίζει, πρέπει να επενδύσετε στο μέλλον του προσωπικού σας. Τέλος, μια πολιτική κινητικότητα του προσωπικού. Δεν είναι σε κανένα οργανισμό καλή ιδέα κάποιος μόλις βγει από το πανεπιστήμιο να προσληφθεί και να περάσει τα επόμενα 40 χρόνια κάθοντας πίσω από το ίδιο γραφείο. Απόκτηση νέων προσόντων, μετακίνηση από πόστο σε πόστο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει πρόγραμμα κινητικότητας που οδηγεί τους ανθρώπους να αλλάζουν θέσεις κάθε 5 με 7 Και γι' αυτό, αυτό αντιβαθάει να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις. Εμείς θα το συνιστούμε αυτό. Σύγχρονος τρόπος για να λειτουργήσετε. Ας έρθουμε τώρα στο θέμα της αντιπολίτευσης και του διαλόγου. Δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε. αλλά πρέπει να αποδίδεται αξία στην αντιπολίτευση. Θα μου πείτε, και γνωρίζω, ο καθένας έχει τα συναισθήματά του μετά το Μαϊντάν, όμως ένα κοινοβούλιο που λειτουργεί σωστά, με μια πιστή αντιπολίτευση, δηλαδή που δείχνει πίστη στο Σύνταγμα, έχει το δικαίωμα να παίξει τον πλήρη της ρόλο. Είναι αντιπολίτευση, δεν είναι πλειοψηφία. Οφείλεται όμως να σέβεστε τα δικαιώματα των εκλεγμένων βουλευτών. Είτε αυτοί βρίσκονται στην πλειοψηφία, είτε συναποτελούν την αντιπολίτευση. Και τουλάχιστον στη διάρκεια τη παρούσα θητεία, το θέμα αυτό δεν έχει αντιμετωπιστεί σωστά. Σα συνιστούμε πολύ θερμά, διότι η πολιτική έχει μόνο μια βεβαιότητα. Όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα, έτσι και εσεί κάποια στιγμή δεν θα είσαστε πλέον ενεργοί βουλευτέ, ή μάλλον θα είσαστε βουλευτέ, αλλά όχι πλέον στην πλειοψηφία θα είστε στη μειοψηφία. Και βασική αρχή του κοινοβουλευτισμού είναι αυτή. Γι' αυτό και θα πρέπει να αποδίδεται αξία στην αντιπολίτευση. Πιστεύουμε ακόμη ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί διακομματικό διάλογο και διαμεσολάβηση. Και εδώ υπάρχουν διάφορα μοντέλα στα διάφορα κοινοβουλευτικά συστήματα και εδώ μπορούμε να σα βοηθήσουμε. Μπορεί να σα βοηθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν και συνεργασίες μεταξύ κομμάτων. Χρειάζεστε όμως και μια γραμματιακή υποστήριξη για να το ενθαρρύνετε και να το υποστηρίξετε αυτό το πράγμα. Είναι καλή ιδέα να συναντάστε, να συνειδριάζετε και διακομματικά, αλλά χρειάζεστε μέθοδο για να στηρίξετε την προσπάθεια αυτή, να την εξυγχρονίσετε και να την θεσμοθετήσετε. Να έρθω στον έβδομο μοχλό, έχει να κάνει με τον ε, κώδικα συμπεριφοράς και την ιδεοντολογία. Κάτι που μας εκπλήσει πάντοτε είναι ότι δεν υπάρχει κάποιος κανονισμός για τον πρόεδρο τον αντιπρόεδρο στη Βουλή όπως ε, με τον τσακωμό που έγινε στη Βουλή κατά τη διάρκεια της επισκέψής μας. Μάλιστα παρακολουθήσαμε περισσότερο από έναν τσακωμούς δεν υπάρχει κανονισμός ο οποίος επιτρέπει λοιπόν στον πρόεδρο να πει ε, θα σας ε, ε αν ε, δεν σταματήσετε. Θα πρέπει να είναι πολύ αυστηρός και ο χρόνος ομιλίας. Θα πρέπει κάθε κοινοβούλιο να ζητά από τα μέλη του και να απαιτεί να γίνεται σεβαστή αξιοπρέπεια του ίδιου του θεσμικού οργάνου. Ιδάλλως να επιβάλλονται κυρώσεις. Σας συστήνουμε λοιπόν να το προβλέψετε αυτό. Υπάρχουν και άλλες συστάσεις, βλέπετε σχετικά, όχι πίσω μου, στο βάθος της αίθουσα, τους κυρίους ε, με τις στολές τους, που είναι οι κλητήρες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εάν ο πρόεδρος πει σε έναν κλητήρια το τάδε μέλος θα ήθελα να αποβληθεί από την αίθουσα και έρθει προς το μέρος σας ο κλητήρας, επιτρέ... Ε, ε, αναμένουμε για λόγους αξιοπρέπειας και σεβασμού και του κλητήρα και του κοινοβουλίου να φύγετε μόνοι σας. Αλλά επίση οι κλητήρε μα φέρνουν τα έγγραφα ή μπορεί να πάνε κάτι από τη μια μεριά τη αίθουσα στην άλλη, προκειμένου να μην υπάρχουν ε, συζητήσει και πηγαδάκια. Ε, χρειάζεται λοιπόν ε, μια ολόκληρη σειρά από μέτρα εδώ. Κάτι που τα περισσότερα κοινοβούλια υιοθετούν. Το άλλο που θα σας συστήναμε και θα μπορούσατε να το δείτε και να καταλήξετε σε έναν κώδικα συμπεριφορά για τη Βερχόπνα Ράντα. Αυτό θα πρέπει να γίνει με τρόπο ανοιχτό και διαφανή. Με διάλογο, με τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών. Έχουμε ένα έγγραφο που, σε αυτό το έγγραφο, μια σειρά από αρχέ που είναι προτάσει για να οργανώσετε βάσει αυτού ένα κώδικα συμπεριφορά και εδώ θα βρείτε και κάποιε αναφορέ σε ιστοτόπου διεθνώ αναγνωρισμένου, όπου υπάρχουν πολλά παραδείγματα κώδικων συμπεριφορά και δοντολογία μπορείτε να το πάρετε και να το προσαρμόσετε στι ανάγκε τη Ουκρανία. Ένα μοντέλο για την Ουκρανία. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε από το μηδέν. Σα το συστήνουμε θερμά. Επόμενη διαφάνεια παρακαλώ. Βάσει των συστάσεων αυτών, την Τετάρτη, την τελευταία ημέρα της εβδομάδας της Ουκρανίας ως προς τις εργασίες μας και τον συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων, και στα πλαίσια τη Συμφωνία Διοικητική Συνεργασία θα υπογραφεί η συμφωνία ακριβώ αυτή μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου από το Γενικό του Γραμματέα και του Γενικού Γραμματέα τη Βερχόφνα Ράντα θα είμαστε συνεργάτες στην μεταμόρφωση της ουρανίας βάσει της συνταγής περισσότερα για περισσότερα. Περισσότερα εσείς θα μεταρρυθμίζετε, περισσότερα εμείς θα σας βοηθούμε για να αξιοποιείτε αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Ε, να σας πω ότι στις αρχές της ιστορίας αυτού του κοινοβουλίου που τότε ονομαζόταν Κοινοβουλευτική Συνέλευση το 1952 και από το 1979 με άμεσες εκλογές ονομάζεται πλέον Ευρωκοινοβούλιο. Σε όλη αυτή λοιπόν την ιστορία δεν υπήρξε ποτέ μια παρόμοια συμφωνία που να έχουμε υπογράψει εμείς με οποιοδήποτε κοινοβούλιο συμπεριλαμβανομένων των κοινοβουλίων των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εν τέλει προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο και αυτό είναι ακόμη μια ένδειξη από τον κύριο Σούλτ, τον κύριο Πλένκοβιτ, τον κύριο Μπρόκ από το Γενικό Γραμματέα ε, ε, της βαθιάς μας αφοσίωσης για να σας ε, στηρίξουμε στην οικοδόμηση δυνατοτήτων στην Περχοφραράντα και γενικότερα στην Ουκρανία. Όλα αυτά θα συμβούν μετά, αργότερα σήμερα, την εβδομάδα αυτή και υπό την αιγύδα του κυρίου Πλέγκοβιτ, τον οποίο αν θέλει μπορεί να σηκωθεί, Ανδρέη. Σε ξέρουν ε, σχεδόν όλοι εδώ, αλλά καλύτερα να σηκωθεί, γιατί κάποιοι από του συναδέλφου τη με κυβερνητική οργανώσει ή κάποιοι από του επισκέπτε μπορεί να μην σε γνωρίζουν. Και επίσης ο, να πω ο ε, ήταν υπεύθυνο και για την ε, αποστολή παρατήρηση στην Ουκρανία και έχει φροντίσει και τις εκθέσεις ε, συνέχειας ε, και συνέχεια της αποστολή αυτή. Είναι πολύ σημαντικές. Η έκθεση αυτή ε, Μάλλον δεν είναι για να φωταγραφηθεί από, με, τα selfies ή από τους φωτογράφους και μετά να την πετάξουμε σε ένα σιρτάρι. Όχι, θέλει να μεταφραστεί σε πραγματικό ενθουσιασμό και να δημιουργηθεί έτσι στη Βερχόφνα Ράντα ένα σύγχρονο, μεταλλαγμένο, δυναμικό θεσμικό όργανο στην καρδιά της Ουκρανικής Δημοκρατίας. Μπορείτε να καταφέρετε κάτι υπέροχο για τη χώρα σας. Και θέλω να σας πω εδώ, ε, εν είδη συμπεράσματος, ότι είχα χθε το βράδυ το προνόμιο να απευθύνω ομιλία προς τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο της Βερχόφνα Ράντα και προς όλους τους αρχηγούς κομμάτων από το Κίεβο. Ε, καθίσαμε γύρω από το ίδιο τραπέζι και ακριβώ αυτή την παρουσίαση του έκανα Είχαμε και ένα πρώτο γύρο συζητήσεων και πραγματικά εντυπωσιάστηκα βαθιά από την προθυμία σε αυτούς τους τόσο δύσκολους καιρούς για, τα πολιτικά πράγματα στο Κίεβο ε, από την αφοσίωση να δείξουν συνεργατική οριμότητα και διάθεση να συνεργαστούν οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, Είχα τόσο κόσμο από το Κίεβ, πρόεδρο και αντιπρόεδρο τη Βουλή, ε, εκπροσώπου των κομμάτων, μέλη τη Φερχοφναράντα και μέλη μη κυβερνητικών οργανώσεων. Carpe diem ήταν το μήνυμα. Αρπάξτε την ευκαιρία και κάντε τα όλα αυτά πράξη. Ξέρετε τι θέλετε να κάνετε. Υπάρχουν οι συστάσεις αυτές και δική σας αποστολή είναι το κοινοβούλιο σας που πρέπει να αναλάβετε την ευθύνη του, το δικό σας σύνταγμα και δική σας χώρα να προχωρήσουν. Εάν συμπλέψουμε σε αυτήν την πορεία πιστεύω ότι θα ε, πετύχουμε κάτι πραγματικά ουσιαστικό καλό για τη χώρα σας. Δεν θα είστε μόνοι σε κανένα μέρος του δρόμου, θα σας συνοδεύουμε σε κάθε βήμα από τους φίλους σας εδώ και όλα τα κοινοβούλια που έχουν αναλάβει συνεργασία μαζί σας, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και διατλαντικός. Και στην τελευταία επίσκεψή μου στο Κίεβο, επειδή τα γνώριζα αυτά, μίλησα εκ μέρου όλων των πρέσβεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, όλων των μελών, αλλά και, με διπλο... εκ μέρου των διπλωματών της, ε, των ΗΠΑ, του Καναδά, τη Ελβετία και τη Νορβηγία. Και αυτό που του έλεγα είναι ότι το βασικό σύνθημα είναι περισσότερα για περισσότερα. Όσα περισσότερα κάνατε, τόσο και εμείς διεθνώ θα αναλαμβάνουμε την ευθύνη να σα στηρίζουμε. Έχουμε δεσμευτεί γι' αυτό και είμαστε καλοί να το καταφέρουμε. Το ίδιο και εσεί. Ευχαριστώ για την Ένα μικρό διάλειμμα τώρα και θα ξαναρχίσουμε στις 4.30 με την επίσημη τελετή έναρξης. Σας έχουν μοιραστεί αυτά. Θα προετοιμάσω τον πρόεδρο Γκρόισμαν και τον κύριο Σούλτ ε, για το έγγραφο αυτό και θα υπάρχει στα Ουκρανικά και στα Αγγλικά στο βάθο τη αίθουσα. Μπορείτε να πάρετε το δικό σα αντίτυπο. Χθε είχαμε τη συζήτηση λοιπόν με του ηγέτε, σήμερα με εσά και αργότερα ξανά με του επίσημου εκπροσώπου για να εργαστούμε σωστά όλη την εβδομάδα, ω την Πέμπτη. Να είμαστε λοιπόν με ενθουσιασμό, με όλε μα τι δυνατότητε και όλη μα την προθυμία και να μην πούμε απλώς ότι θα κάνουμε κάτι, αλλά να το μεταφράσουμε σε πράξη.